Ίας έμπολα. Εξ του Συμβουλίου. Ο Ιταλός Υπουργός. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κύριε Επίτροπε. Η πρόσφατη επιδημία του έμπολα στη Δυτική Αφρική είναι η πιο σημαντική στο είδος της. Είναι μια υγειονομική δημόσια επίγουσα κατάσταση που δημιουργεί τεράστιες διεθνεί ανησυχίε. Η επιδημία του έμπολα έχει τρομακτικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και σε ανθρωπιστικό επίπεδο σε χώρες που έχουν πληγεί και σε όλη την περιοχή της Αφρική. Το Συμβούλιο είναι πάρα πολύ ανήσυχο για τις ε, συνέπειες σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και την ασφάλεια των χωρών της Δυτικής Αφρικής που έχουν πληγεί από το έμπολα. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι το, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη των Ασθενειών ε, εκτιμάει ότι μπορούν να αρρωστήσουν από το έμπολα και οι ε, πίκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν εκεί. Αλλά αν όμως ακολουθήσουν τις συστάσεις ε, δεν κινδυνεύουν. Εμείς μαζί με την διεθνή κοινότητα θέλουμε να αντιδράσουμε στην επιδημία. Ε, στις 15 Αυγούστου οι Υπουργοί Εξωτερικών προσπάθησαν να συντονίσουν ούτως ώστε να υπάρξει διεθνής οργανωμένη απάντηση. Και στις, ε, στις 30 Αυγούστου το έκτακτο συμβούλιο μίλησε για τη σημασία να υπάρξει μια διεθνής υποστήριξη συντονισμένη το συντομότερο δυνατόν και όσο πιο αποτελεσματική. Ζήτησε μέγιστο συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και κάλεσε το Συμβούλιο να υιοθετήσει ένα πλαίσιο συνολική απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ποιε ήταν οι παρεμβάσει μα επίπεδου follow-up για το έμπολα. Σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αντέδρασαν στην ε, κρίση του έμπολα από την αρχή. Αυτό σημαίνει υποστήριξη οικονομική στις οργανώσεις των γιατρών, του ΟΗΕ, της ανθρωπιστικές. Ε, βοηθάμε τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και ορισμένοι ε, πλήρωσαν αυτή τη δέσμευση με τη ζωή τους. Ε, ο στενός συντονισμός με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για να γίνουν κοινέ αναλύσεις για να εκτιμήσουμε την ανάγκη για ανθρωπιστική παρέμβαση. Ο μηχανισμός αστικής προστασίας ενεργοποιήθηκε κατόπιν αίτησης του, της Διεθνής Οργάνωσης Υγείας το κέντρο συντονισμού το, της απάντησης ε, επίγουσας ε, είναι λειτουργικό ε, κάθε μέρα, κάθε ώρα και συντονίζει τη βοήθεια. Από την επιδείνωση της κρίσης τα κράτη-μέλη πέτειναν την υποστήριξή τους και έδειξαν διάθεση να προσκομίσουν περαιτέρω βοήθεια και ιατρικό προσωπικό. Θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα πολύ γρήγορα. Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε ε, δημιουργώντας ένα κέντρο για να βοηθήσει τους πληγέντες στην Σιέρα Λεόνε που θα είναι ε, σύντομα ε, λειτουργικό. Η Αυστρία και η Γαλλία έδωσαν υλικό σε είδος, ιατρικό υλικό κτλ. Η Γερμανία βοηθάει επίσης, η Ιταλία βοηθάει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από την αρχή της κρίσης και έδωσε και 200 εκατομμύρια ευρώ για τις δραστηριότητες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ε, στην Κινέα. Ακόμα 240.000 ευρώ ε, θα δοθούν σύντομα. Επίσης, ε, εγκρίναμε μία παρέμβαση για 1,2 εκατομμύρια ευρώ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ιού. Το Συμβούλιο ετοιμάζει μια παγκόσμια απάντηση, μια συνολική απάντηση Ευρωπαϊκή Ένωση για την κρίση. Και θα προωθήσουμε το συντονισμό των αέριων μεταφορών, ε, που είναι ένα σημαντικό κενό αυτή τη στιγμή και περιορίζουν την πρόσβαση του ιατρικού προσωπικού και ανθρωπιστικού προσωπικού στην ε, περιοχή, καθώ και του ιατρικού υλικού. Βεβαίω γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την ανάγκη να κάνουμε περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει ούτω ώστε να επανοικοδομηθούν, επανοικοδομηθούν τα ιατρικά συστήματα που έχουν καταρρεύσει λόγω του έμπολα. Αν δεν το κάνουμε, η ανθρωπιστική κρίση του έμπολα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλε χώρε τη Αφρικανική Υπήρου. Η Προεδρία μαζί με την ε, Κομισιόν θα συντονίσει την ε, συλλογική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εταιρική σχέση με τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είμαστε ενεργοί σε πλαίσιο, στο επίπεδο της ε, δημόσιας υγείας για να υποστηρίξουμε και, τις, και τη ζωή, την ανθρώπινη ζωή των υπηκόων μας. Ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με την Κομισιόν συντονίζουν τις αποκρίσεις τους στις μεγάλες απειλές για την ε, υγεία μαζί με την ε, Επιτροπή για την Ασφάλεια της Υγείας. Διάφοροι φορείς, η Κομισιόν και το Κέντρο για την Πρόληψη των Ασθενειών είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία την επιδημιολογική των μεταδοτικών ασθενειών και τα υγειονομικά προβλήματα που συνδέονται. Ε, έγινε στις Βρυξέλλες το Σεπτέμβριο μια συνεδρίαση υψηλού επίπεδου για να συντονίσουμε τις περαιτέρω φάσεις της απάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιδημία του έμπολα στη Δυτική Αφρική. Πέρα από τους αρμόδιους ε, επιτρόπους, τους διάφορους υπουργούς υγείας των κρατών μελών, στη συνεδρίαση συμμετείχαν ως συντονιστής υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ για την για τον ιό του έμπολα, καθώς και εκπρόσωποι των Διεθνών Οργανώσεων Υγείας, μη κυβερνητικών οργανώσεων και των γιατρών χωρίς σύνορα. Η συνεδρίαση ήταν η αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας συντονισμού της διεθνούς απόκρισης που είναι απαραίτητη για να καταπολεμήσουμε την επιδημία. Οι Υπουργοί Υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν το θέμα στη συνεδρίαση την Υπουργική, την άτυπη που θα γίνει στο Μιλάνο στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου και θα μιλήσουν ειδικά για τις ε, επικείμενες δράσεις, ε, το follow-up, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ε, τα ταξίδια των Ευρωπαίων υπηκών, η ανάγκη να επιμεριστούν οι πόροι για να αντιμετωπίσουμε τις επίκουσες καταστάσεις, να δώσουμε στη διάθεση της Αφρικής εμβόλια κατά του ιού, να υποστηρίξουμε τις πληγήσεις χώρες, τους μη κυβερνητικού οργανισμούς, τον ΟΗΕ και τα λοιπά, όλους όσους είναι ενεργοί στην περιοχή, ούτω ώστε να ενισχύσουμε την, το συντονισμό ε, που κάνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο ΙΕ. Ε, αγαπητοί βουλευτές, κυρία Επίτροπε, ήμουν αρκετά αναλυτικός για να λάβω υπόψη και να σας εξηγήσω την δέσμευση που έχει λάβει το Συμβούλιο για να βοηθήσει τις πληγήσεις χώρες και τις διεθνείς οργανώσεις στην καταπολέμηση, στον αγώνα κατά της τεράστιας αυτής επιδημίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Επίτροπος Γεωργίευα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία πλήρη παρουσίαση από το Συμβούλιο ακούσαμε. Αυτό που θα ήθελα εγώ να κάνω είναι να συνεισφέρω σε αυτή τη συζήτηση υπησερχόμενη περισσότερο σε τρία σημεία. Πρώτον, τον χαρακτήρα αυτής της επιδημίας Δεύτερον, τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει μια συντονισμένη απάντηση σε αυτή την επιδημία. Και τέλος κάποια λόγια για την δυνατότητα να προστατέψουμε τους ίδιους τους πολίτες της Ευρώπης μέσα από τη δράση μας. Για την ίδια την επιδημία της έμπολα. Είναι κάτι χωρίς προηγούμενο, διτά, με δύο τρόπους. Πρώτον, επειδή είναι μια πανδημία και επειδή συμβαίνει σε χώρες με πολύ αποδυναμωμένα, αδύναμα συστήματα υγείας ως πρώτη παρατήρηση. Σε τέτοιου είδους πανδημίες στο παρελθόν ήταν σε μέσου εισοδήματος χώρες όπου υπήρχε η δυνατότητα να κινητοποιηθεί η σωστή απάντηση στις χώρες αυτές. Τώρα δεν είναι δυνατόν αυτό σε αυτές τις φτωχές χώρες. Και δεύτερον, σε σχέση με τέτοιου είδους επιδημίες δεν υπήρξε τέτοια διάρκεια όπως αυτή της πανδημίας της έμπολα τώρα και που διαρκεί τόσο πολύ. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά πολύ δραματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και όπως αναφέρθηκε από πλευράς του συντονιστού του των Ηνωμένων Εθνών του δόκτωρα Ντέιβιντ Ναβάρο εξαιρετικά ε, σοβαρού επιστήμονα και που βλέπουμε ότι έχουμε χιλιάδες περιπτώσεις ε, και μάλιστα με ε, ελάχιστα, με πολύ, λίγα, με πολύ λίγες κλίνες. Όμως το πιο ανησυχητικό στοιχείο το οποίο βλέπουμε είναι ο διπλασιασμός περίπου του αριθμού των ε, ασθενών κάθε τρεις εβδομάδες και αν δεν δράσουμε με αποφασιστικότητα τώρα υπάρχουν τρεις μεγαλύτεροι, μεγάλοι κίνδυνοι που απορρέουν. Πρώτον, σε αυτές τις τρεις χώρες, ε, Γουινέα, ε, Σιέρα Λεόν ε, και Λιβερία να μπορέσει να διαδοθεί η νόσος αυτή και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναχαιτιστεί είναι ήδη δύσκολο να αναχαιτιστεί σήμερα θα είναι πολύ πιο δύσκολο στο μέλλον δεύτερο μπορεί να μην είμαστε σε θέση να προστατέψουμε άλλες χώρες σε αυτή την περιοχή από την διάδοση αυτής της ε, ε, πανδημίας και μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις ακόμα και το τρίτο και το πιο επικίνδυνο ως κίνδυνος είναι όσο περισσότερο δεν καταφέρνουμε να ελέγξουμε την κατάσταση κατάσταση τόσο μεγαλύτερη, μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να βρεθεί εκτός ελέγχου αυτός ο, ο ιός και είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να λάβει δραματικές διαστάσεις. Δεν κάνουμε πια λόγο απλά το, να βοηθήσουμε με έκτακτα μέτρα ε, κατεπήγοντος χαρακτήρα σε αυτές τις τρεις χώρες βλέπουμε ότι υπάρχει επίπτωση στις οικονομίες τους και στις κοινωνίες τους που είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι επιπτώσεις. Ανησυχούμε και για τις πολιτικές ε, ε, επιπτώσεις ε, και τις επιπτώσεις όσον αφορά την ασφάλεια σε αυτές τις χώρες. Είναι χώρες που βίωσαν εμφυλίους πολέμους κατά το παρελθόν. Μόλις άρχισαν να ανοικοδομούν τις κοινωνίες τους και τώρα με αυτόν τον τρόπο πλήττονται με ιδιαίτερο τρόπο πάλι. Και όταν βλέπουμε την, ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η έμπολα στο, στην πρώτη γραμμή του μετόπου, να κινητοποιήσουμε ανθρωπιστική βοήθεια, να αποσταλούν εκεί τα στελέχη, να βοηθήσουν επιτόπου. Απαιτούνται υψηλή ε, παιδείας και κατάρτισης άτομα ως στελέχη. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με στελέχη, εξοπλισμό και θέματα μεταφοράς. Υπησέρχομαι στο δεύτερο σημείο. Τι κάνουμε από πλευρά Ευρώπη, ώστε στην πρώτη γραμμή του μετόπου να καταπολεμήσουμε την έμπολα. Φυσικά κινητοποιούμε κονδύλια, χρήματα. Και είμαι υπερήφανη που μπορώ να πω ότι η Επιτροπή με 150 εκατομμύρια ευρώ που κινητοποιεί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εκείνων που χορηγούν για να υπάρξει συνεισφορά στην αντίδρασή μας, στη δραστηριοποίησή μας κατά της κρίσης αυτής θα διασφαλιστούν τα κονδύλια που είναι αναγκαία. Αυτό που κάνουμε είναι διασφαλίζουμε τα κονδύλια και θα κάνουμε και ακόμα περισσότερα. Τα κράτη-μέλη μας τη Δευτέρα μέχρι 78 εκατομμύρια ευρώ υποσχέθηκαν θα δεσμεύσουν. Και πολλοί προσπαθούν να αυξήσουν την χρηματοοικονομική του συνεισφορά ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο μέλλον. Πολύ πιο σημαντικό από τα χρήματα είναι να κινητοποιήσουμε την αρρωγή και βοήθεια επιτόπου με πειραματικά εργαστήρια που δημιουργούνται και υπάρχουν σε αυτά τα κράτη και συνεισφέρουν τα κράτη-μέλη ώστε να υπάρξουν νέες κλινικές, νέα νοσοκομεία για να διασφαλιστούν οι αναγκαίε κλίνες για τους ασθενείς να σας πω σε σχέση με τους ε, αριθμούς όταν ε, αναφέρεται ότι στις ε, εκατοντάδες οι επιδόσεις είναι καλό αυτό αλλά χρειάζονται χιλιάδες χιλιάδες όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία αποστέλλονται σε αυτές τις, από αυτές τις κοινότητες ως ασθενείς με όλους τους κινδύνους προσπαθούμε να δράσουμε σε αυτό το κρίσιμη σημασία σημείο που είναι η εκένωση από πλευράς ιατρικού, ιατρικής δράσης. Τι θα μπορέσουμε να κάνουμε αν κάποιος έχει μολυνθεί, πώς θα μπορέσει να βοηθηθεί άμεσα. Στην Ευρώπη προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την δυνατότητα ε, κένωσης ε, και αποκλεισμού των ε, όσων έχουν μολυνθεί ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν από ιατρικής πλευράς άμεσα. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, κατανοούμε την κρίσιμη σημασία στο να υπάρξουν επενδύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη, για τα εμβόλια, για την δυνατότητα της αντιμετώπισης αυτού του ιού, της έμπολα. Και υπήρξε και συζήτηση εδώ στην Ευρωβουλή όσον αφορά και τον, ε, ε, την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, για αυτά τα θέματα. Υπησέρχομαι στο τρίτο τώρα σημείο, το οποίο είναι τι κάνουμε για την ασφάλεια των δικών μας πολιτών στην Ευρώπη. Πήραμε το, μήνυμα το οποίο ήταν σαφέστατο και ε, ευκρινέστατο. Να πω δύο πράγματα. Πρώτον, εμείς αυτό που λέμε είναι να σταματήσει αυτός ο ιός εκεί που βρίσκεται, να απομονωθεί. Να απομονωθεί και να δράσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ας μην απομονωθούν όμως οι χώρες. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στην Brussels Airlines, στην Air France, ευρωπαϊκές ε, εταιρείες εναέριων μεταφορών που εξακολουθούν να δρουν στις μεταφορές πρώτα και από αυτές τις χώρες. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Δεν θα ε, μπορέσει να διεισδύσει αυτός ο ιός στην Ευρώπη και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή τεράστιο έργο επιτελείται για να διασφαλίσουμε ότι το πειραματικό μας δίκτυο των πειραματικών μας ε, δυνατοτήτων θα είναι επαρκές. Να έχουμε την σωστή ε, θεραπεία που θα προσφέρεται, να συντονίζουμε τα μέτρα πρόληψης από πλευράς μας και να μπορούμε με μια φωνή να συνεννοούμαστε και να ενημερώνουμε και να επικοινωνούμε. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι με ενεθάρρυνε ιδιαίτερα η συνάντηση της Δευτέρας. Η Ευρώπη πραγματικά δρά ως ένα, ένας ενιαίος φορέας. Παρακαλώ, οι συντονιστές, πρέπει να δράσουμε όλοι με συντονισμένο τρόπο και από κοινού θα τα καταφέρουμε έτσι. Ευχαριστώ. Δύο λεφτά, Στύρπερ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και η Επίτροπος, κυρία Πρόεδρε, αυτός ο ιός εξαπλώνεται με πραγματικά εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Αν ακούσουμε τα στοιχεία που έχει στείλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μπορεί ε, να φτάσουμε και τα 20.000 κρούσματα ε, ε, μετά τα Χριστούγεννα. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση με ε, σοβαρότητα και όχι με στόχο τον εντυπωσιασμό. Δεν θα πρέπει να πέσουμε θύματα του πανικού, αλλά θα πρέπει να βροντοφωνάξουμε πως η διεθνή κοινότητα υποεκτίμησε την επιδημία του ιού ε, έμπολα και το μήνυμα που θα στείλουμε θα πρέπει να είναι σαφής. Η κρίση με τον έμπολα δεν είναι μόνο πρόβλημα για τη Δυτική Αφρική, είναι μια απειλή παγκόσμια. Χρειάζεται λοιπόν μια αποφασιστική απόκριση ήδη σήμερα και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τα όσα έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Είναι βήματα πολύ σημαντικά, αλλά δεν είναι αρκετά. Οι δικές μας οργανώσεις και θα πρέπει οι απεσταλμένοι μας επιτόπου να εισακουστούν γιατί είπαμε ότι χρειάζονται όχι τόσο πολύ χρήματα όσο οργάνωση, ανθρώπινη πόροι, βοήθεια σε τεχνολογικό ε, επίπεδο, όπως επίσης και η ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Αυτή τη στιγμή υπολείπονται πολύ οι δομές υγείας ε, στην Αφρική και δεν υπάρχει και αρκετό υγειονομικό προσωπικό. Και τι είναι το πιο σημαντικό. Θα πρέπει να ενημερώνεται ο ντόπιο πληθυσμό. Δεν είναι αρκετά ενημερωμένο και γι' αυτό θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διπλασιάσει τι προσπάθειε που κάνει. Ξέρουμε πως ε, θα συναντηθούν οι Υπουργοί Υγείας στο Μιλάνο, άτυπα. Θα πρέπει να μας παρουσιάσουν ένα επίγον σχέδιο δράσης έτσι ώστε να σταθούμε δίπλα στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δράσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φανεί γενναιόδορη. Όχι μόνο να είμαστε αλληλέγγυοι ε, προς τη Δυτική Αφρική, αλλά για να εξασφαλίσουμε πως θα είναι ασφαλείς και οι δικοί μας πολίτες. Ο χρόνος πιέζει και η ε, απόκριση που θα δώσουμε θα πρέπει να είναι αποφασιστική. Δύο λεφτά, κυρία Μακάβαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο που μας παρουσίασαν σήμερα τα βήματα που λήφθησαν τούτη την εβδομάδα, που είναι η κρίσιμη εβδομάδα για να το αντιμετωπίσουμε. Μιλήσατε για το Παγκόσμιο Οργανισμό ε, υγείας ε, συνάδελφα και είπατε πως 20.000 κρούσματα, 20.000 θάνατοι πριν ή μετά τα Χριστούγεννα. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως θα πρέπει οι προσπάθειές μας να επιταχυνθούν, να κάνουμε περισσότερα. Ε, τα όσα έγιναν τη Δευτέρα στην, στην Βρυξέλλες με ικανοποίησαν ιδιαίτερα, όπως επίσης και ανακοινώσει του Προέδρου των ΗΠΑ που ακούσαμε θα λάβει ε, πλέον ε, ε, μέρος στις προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για να καταπολεμηθεί ο έμπολα. Χρειαζόμαστε λοιπόν και πρόθεσμα μέτρα, δηλαδή έλεγχος επιτόπου δράση και παράλληλα να δούμε σε μακροπρόθεσμο επίπεδο τι θα καταφέρουμε, γιατί ξέρουμε πως όλοι καθυστερήσαμε να αντιδράσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε γιατί η επιδημία αυτή είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι οποτεδήποτε στο παρελθόν. Γιατί είχαμε περισσότερους θανάτους τώρα από τότε, έχουμε τους περισσότερους θανάτους σήμερα από τότε που εντοπίστηκε πριν από 40 χρόνια αυτή η ασθένεια. Γιατί τα εμβόλια και οι θεραπείε ε, δεν ε, έχουν ε, βγει στην αγορά, γιατί έχουμε πειραματικά εμβόλια που δεν έχουν φέρει τα αποτελέσματα που επιθυμούμε, για να είμαστε σίγουροι πω την επόμενη φορά θα κάνουμε τι ερευνητικέ προσπάθειε και ακόμα και όταν πάψουμε να είμαστε στα πρωτοσέλιδα, οι έρευνε αυτέ θα συνεχιστούν. Ξεκίνησε η δοκιμή, η πραγματική δοκιμή ενό φαρμάκου σήμερα στι ΗΠΑ και ελπίζω πω αυτή αυτή η νοσοκομιακή δοκιμή θα οδηγήσει σε εμβόλιο που θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Και τέλος να αποτίσω ένα φόρο τιμής στους υγειονομικό προσωπικό ε, και στους γιατρούς που βρίσκονται επί τόπου από τα κράτη-μέλη αλλά επίσης και σε όλους τους ε, ομολόγους τους από την Αφρική οι οποίοι είναι πολύ γενναίοι και οι οποίοι με πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας κάνουν ό,τι μπορούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είπε, θα πρέπει να ενισχύσουμε τα συστήματα υγείας στις χώρες αυτές και αν αναλάβουμε αυτή τη δέσμευση τότε Οπότε αυτή είναι και μια καλή επένδυση για τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί έτσι προστατευόμαστε και εμείς στο εσωτερικό των χωρών μας. Άρα λοιπόν, βραχυπρόθεσμα έλεγχος, μακροπρόθεσμα περισσότερο προβληματισμό για το θέμα τούτο. Mr. Deva, you have the floor for one minute. Ο κύριος Ντέβα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με θαρρύνουν όλα αυτά που είπε η Επίτροπος Γεωργίευα για όλα όσα κάνουμε θα πρέπει να ξεκινήσουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, καθώς εξαπλώνεται ο ιός, ε, εξαπλώνεται και μέσω του μολυσμένου κρέατος, του κρέατος που καταναλώνει ο κόσμος. Θα πρέπει να περιορίσουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση να εμπλακούν σε αυτό το πρόγραμμα περιορισμού. Θα πρέπει ε, τα μεγαλύτερα κράτη της Αφρικής να βοηθήσουν τα πιο αδύναμα κράτη της Αφρικής γιατί είναι πρόβλημά τους αλλά και δικό μας πρόβλημα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, διακινδυνεύουν τη ζωή τους από το ιατρικό προσωπικό για να σώσουν ζωές. Θέλω επίσης να, ζητήσω, να ρωτήσω την ε, Επίτροπο αν υπάρχει εμβόλιο αυτό που έχουν στις ΗΠΑ μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία ε, και να μην περιμένουμε μέχρι να επιταθεί η κρίση και έχουμε περισσότερους θανάτους. Ο κύριος Γκέρνης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Υποεκτιμήσαμε στη διεθνή κοινότητα την κρίση και δεν είχαμε και καλά συντονισμένη στρατηγική. Και αυτό εξηγεί γιατί τόσο ανησυχητικά εξαπλώθηκε ο ιός. Η απόκριση είναι, στο κάναμε αρκετά είναι όχι. Ο αριθμός κροσμάτων διπλασιάζεται κάθε δύο εβδομάδες. Όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο πιο πολύ θα εξαπλωθεί. Θα πρέπει λοιπόν για τον έβολα εμείς να ε, εργαστούμε με πολλαπλάσιους ρυθμούς. Και τι σημαίνει αυτό. Προφύλαξη. Θα πρέπει στα μίντια ε, να καταφέρουμε ε, να ενημερώσουμε τον πληθυσμό έτσι ώστε και να μην εξαπλωθεί εκτός των απομονωμένων ε, περιοχών ο ιός αλλά και να ενημερωθεί καλύτερα ο κόσμος για τι πρέπει να κάνει. Ξέρετε πως όλοι οι μεγάλοι ανθρωπιστές μίλησαν για το τι πρέπει να κάνουμε. Μία έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για να κινητοποιηθούν όλα τα μέσα, ακόμα και τα στρατιωτικά, και να χρησιμοποιηθούν υπό τη διεύθυνση των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι αυτό πλέον θα πρέπει να ξεφύγει από τη σφαίρα των λόγων και να περάσουμε στη δράση. Πρέπει σε όσου έχουν μολυνθεί να προσφέρουμε θεραπείες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι δομές. Πολύ συχνά τους ασθενείς του ε, τους πετάνε έξω από τα νοσοκομεία, τα οποία έχουν ε, γεμίσει από ασθενεί, γιατί περιμένουν να αφήσουν τα νέα κρούσματα ε, να έρθουν ε, όπως για παράδειγμα στη Λιβερία όπου δεν υπάρχει σύστημα υγείας που να μπορεί να φροντίσει τέτοιο μεγάλο ρυθμό ασθενών. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε πως η δική μας ε, απόκριση δεν ήταν αρκετή γιατί το πρόβλημα είναι τέτοιο που ενδεχομένως να καταρρεύσουν και τα συστήματα υγείας των όμορων περιεχών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τις ε, χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή απειλούνται μπορεί να καταρρεύσει και η βιομηχανική τους και η αγροτική τους ε, περιοχή με αποτέλεσμα να χρειάζονται όλο και περισσότερο ανθρωπιστική βοήθεια και ένας φόρος όσοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους εκεί. Ο κύριος Σάντσες, μισή λεπτό παρακαλώ. Η κυρία Σάντσες, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ξέρουμε πώς είναι οι νεκροί από αυτή την πανδημία της έμπολα. Τα συστήματα υγείας της Δυτικής Αφρικής είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και έχουν καταρρεύσει, καταρρεύσει τώρα. Δύο γιατροί ανά χίλιου κατοίκους για να αντιμετωπιστεί αυτή η χωρίς προηγούμενο πανδημία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαντάζονται τίποτα άλλο παρά να περικοπεί ε, η βοήθεια στην ανάπτυξη στα κονδύλια της. Και βλέπουμε αυτό σε σχέση με το 2011 τι σημαίνει. Δεν είναι φιλανθρωπία η ελεημοσύνη, είναι δικαιοσύνη η βοήθεια για την ανάπτυξη και έχουμε τεράστιο χρέος για τις αφρικανικές χώρες ε, και για τους πόρους ε, σε σχέση με την Αφρική. Φαίνεται ωστόσο ότι οι χώρες του Νότου δεν μπορούν να τύχουν προτεραιότητας. Πρέπει όμως να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου αυτή η απειλή που βρίσκεται σε παγκόσμιο επίπεδο να μας κινητοποιήσει για να γίνει κάτι από πλευράς μας. Επιπλέον σε σχέση με την Ευρώπη για την κινητοποίηση τη υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν ε, ε, αντιδρά όπως πρέπει. Χρειάζονται ιατροί, πειραματικά εργαστήρια, δυνατότητες απομόνωσης των όσων έχουν μολυνθεί. Δεν, δεν χρειάζεται στρατιωτική υποστήριξη. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Κούβας ε, που εκατοντάδες γιατρούς αποστέλει ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και όχι αυτό που κάνουν οι ΙΠΑ αποστέλλοντας χιλιάδες στρατιώτες ε, περισσότεροι στρατιώτες από ότι γιατροί ή ε, ιατρικό προσωπικό. Και πρέπει εδώ να μην στρατιωτικοποιηθεί περισσότερο αυτή η περιοχή του κόσμου. Είναι κατεπήγον να υπάρξει ένα πρόγραμμα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε κατεπηγόντω να κινητοποιηθεί η Ευρώπη υπέρ τη ε, ε περίθαλψη και τη ιατρική βοήθεια. Δεν μπορούμε να αναμένουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Ριβάζει 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθουμε λιγάκι στον τρόπο διαχείρισης και κακής διαχείρισης αυτής της επιδημίας. Κοιτάξτε, ξεκίνησε στις 22 Μαρτίου στην ε, Γινέα. Πήγε στην ε, Σιαραλεόνε, στη Λιβερία, τώρα στη Σενεγάλη και στην Ιγυρία. Και όπως είπατε, υπάρχουν πάνω από 4.900 άτομα. Αλλά αυτή είναι μια εκτίμηση, γιατί δεν ξέρουμε πόσοι έχουν μολυνθεί. Πάνω από 2.500 νεκροί. Η διεθνής κοινότητα ούτε δεν αντέδρασε γρήγορα ούτε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία. Λένε θα κάνουμε αυτά που κάνουμε συνήθω. Θα περιορίσουμε την επιδημία, αλλά τελικά αναπτύσσεται εκθετικά. Ξέρουμε ότι οι χώρε δεν μπόρεσαν να αποκριθούν. Ε, γιατί πρόκειται για μια κατάσταση πολέμου. Όταν βλέπουμε την κατάσταση στη, Λιβ... στη Λιβυρία, λέει ο Πρωθυπουργό, θα καταρρεύσει η χώρα μου. Δεν υπάρχει υγειονομικό σύστημα, δεν υπάρχει ε, επιχειρηματικότητα. Υπάρχει και το φάσμα τη διατροφική ασφάλεια. Όταν η Κομισιόν λέει έχουμε 150 ε, εκατομμύρια ευρώ να δώσουμε. Δεν αρκούν. Υπάρχει έλλειψη διεθνού συντονισμού. Εμείς θα θέλαμε ο ΙΕ μέσω του ΟΤΣΑ για την ανθρωπιστική βοήθεια να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Γιατί χρειάζεται πραγματικό συντονισμό. Όταν ακούω τον πρόεδρο Ομπάμα να λέει ε, θα στείλουμε 3.000 στρατιωτικού Θέλω να απαντήσω στον συνάδελφο. Δεν είναι 3.000 στρατιωτικοί, είναι 3.000 άτομα τα οποία θα δημιουργήσουν νοσοκομεία. Νοσοκομεία για να ανταποκριθούν στην ανάγκη που υπάρχει. Αλλά κυρίε και κύριοι, δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει η Κομισιόν να πει, ένα και εμεί θα βοηθήσουμε για να στηθούν νοσοκομεία, και εμεί θα στείλουμε προσωπικό. Εγώ έχω τους, τα παιδιά μου που είναι γιατροί χωρί σύνορα εκεί πέρα, αλλά η κατάσταση είναι καταστροφική. Όταν ακούω τον Επίτροπο Μπόρκ να λέει Α, ο κίνδυνο είναι χαμηλό στην Ευρώπη. Δεν έχει καταλάβει τίποτα αυτό ο κύριο. Αν μεταλλαχθεί αυτό ο ιό, θα γίνει παγκόσμια επιδημία. Καταλαβαίνετε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εύρο του προβλήματο. Και τελευταίο που θέλω να σα πω. Πολύ ωραία που λέμε. Ναι, πρέπει να επαναπατρίσουμε κάποια άτομα. Χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Αλλά ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα αεροπλάνο που να μπορεί να επαναπατρίσει κάποιον εθελοντή. Και σκεφτείτε όλου αυτού τι ανθρωπιστικέ οργανώσει που δουλεύουν εκεί. Κοράω για δύο λεφτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η επιδημία έμπολα στην Βόρεια Αφρική έχει τεράστια επίπτωση σε υγειονομικό επίπεδο και τρομερό κόστο σε ανθρώπινε ζωέ πάνω από 2.500 νεκροί και περίπου 5.000 συμμολυσμένοι. Στις ε, αφρικανικές χώρες που έχουν πληγεί κυρίως από τον, ιό δεν έχουμε εγγύψει επαρκώς. Εμείς ανησυχούμε και κινητοποιούμαστε. Εντάξει. Κάθε φορά βέβαια που μολύνεται ένας δυτικός υπήκος. Αλλά την ίδια ε, πρεμούρα, την ίδια, το ίδιο πάθος, την ίδια αγωνία δεν την έχουμε όταν ε, πλήττονται εκατομμύρια θύματα ε, στην Αφρική, την έχουμε την Αφρική μόνο για να την εκμεταλλευόμαστε, έτσι. Ποια είναι η καλύτερη ευκαιρία από αυτή την επιδημία του έμπολα για να αρχίσουμε και εμείς να ανασκουμπωνόμαστε, να ανασκουμπώνονται και οι πολυεθνικές οι οποίες ε, ε, δρέπουν τόσους καρπούς από την Αφρική, ε, γδίνοντας από τους πόρους τους. Η Αφρική δεν είναι μόνο θάνατη, φόβος, μόλυνση κτλ. Είναι και κοινωνικονομικά προβλήματα, τρομερά. Ο ΦΑΟ πριν από λίγο μίλησε για το τεράστιο πρόβλημα με τις οδιές στην ε, Βόρεια Αφρική. Ε, τα προβλήματα της κρίσης είναι όλο και πιο έντονα ε, και πλήττεται η όλο και πιο ασθενής οικονομία των χωρών αυτών. Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι τρομακτική οι τοπικέ αρχέ και, οι θεσμοί δεν αρκούν. Ε, τα υγειονομικά συστήματα είναι ασθενή ε, και μερικέ φορέ δεν υπάρχουν καν. Δεν υπάρχουν ε, βασικέ υποδομές, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν απαραίτητε δομέ για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει μια τελείω στρεβλή εικόνα για την αρρώστια από, από τις τοπικές κοινότητες, γιατί καταρχάς είναι και αναλφάβητη και αυτό βοηθάει την εξαρτήση του ιού. Υπάρχουν ε, τρομερές, τρομερά προβλήματα, συγκρούσεις εντάσεις ας πούμε σε επίπεδο εθνοτήτων, κοινοτήτων κτλ. που αυξάνουν τους νεκρούς. Το ερώτημά μου συνάδελφοι είναι η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες τρομακτικές προκλήσεις και αν ναι με ποιο τρόπο. Σαλβίνη, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς. Και η Ευρώπη ξυπνάει τελευταία και καθιδρωμένη. Μιλάμε για έναν ιό που ε, έχει χρόνο επόασης από 2 μέχρι 21 μέρες. Ε, εμείς έχουμε το, τη, λεγόμενη την επιχείρηση Mare Nostrum για να αντιμετωπίσουμε τις ε, βάρκες ε, με τους μετανάστες από Νιγηρία, από τη Σενεγάλη, από Λιβερία, από τις χώρες που πλήγονται κιόλας από τον ιό. Ε, όσο πιο γρήγορα ξυπνήσουμε, τόσο καλύτερα για όλους μας και κυρίως ε, για αυτούς ε, τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή στις, ε, στα δελτία ειδήσεών μας. Έχουμε. Η Σαουδική Αραβία και η Κορέα σκέφτονται να κλείσουν τα σύνορα στους μετανάστες που προέρχονται από αυτές τις περιοχές. Εμείς τι κάνουμε, πέρα από το να πηγαίνουμε εκεί για να σώσουμε ζωές και το κάνουμε και καθυστερημένα, έτσι, για να αποφύγουμε τα προβλήματα εδώ. Λοιπόν, σας ρωτάω, η Ευρώπη μπορεί να το παίζει ότι δεν τρέχει τίποτα όταν ξεμπαρκάρουν εδώ χιλιάδες άτομα που πέρα από τον ιό έμπολα μπορεί να είναι και φορείς και είναι και φορείς. Αυτά λένε ε, και τα Ιταλικά μέσα ενημέρωση, φυματίωση και άλλου ιού και δεν σταματάει εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ιταλικό, είναι ευρωπαϊκό. Έχει νόημα να πηγαίνουμε εκεί για να πιάνουμε αυτά τα άτομα από τη θάλασσα χωρίς καμία ε, εγγύηση ή μήπως τα λεφτά που ξοδεύουμε για το Mare Nostrum θα τα καλύτερα να τα ξοδέψουμε στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική για να σταματήσουν αυτοί, αυτά τα ταξίδια του θανάτου και να, για να αποφύγουμε στα παιδιά μας το φάσμα της μόλυνσης. Βέντα. 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε στην Δυτική Αφρική βιώνουμε την περίπτωση της έκρηξης του ιού έμπολα. Είχαμε ε, κάποιες εκατοντάδες ε, περιπτώσεις ε, και χιλιάδες ε, ε, που μολύνθηκαν και ε, αποβίωσαν. Επίσης από πλευράς ιατρικού προσωπικού υπήρξαν θύματα. Δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές, επαρκείς υποδομές για να βοηθηθούν οι ασθενείς. Δεν υπάρχουν αρκετές γνώσεις καν για αυτή την ασθένεια εκεί. Αυτή η πανδημία έχει διεθνείς διαστάσεις είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και μπορεί να καταλήξει και στην Ευρώπη στο τέλος τέλος και να πλήξει τους πάντες. Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι Αφρικανοί, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια ώστε να προλάβουμε άλλες ε, πανδημίες. Ε, το ψήφισμα είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο έχουμε καταθέσει. Υποστηρίζουμε τα 140 εκατομμύρια ε, βοήθειας στις χώρες που έχουν πληγεί. Είναι πολύ σημαντικό να καταπολεμηθεί ο ιός και σε σχέση με τον, την αύξηση του αριθμού των ε, θυμάτων ε, είναι πραγματικά κάτι ε, κατεπήγον. Μόνο με τη βοήθεια των ε, Ευρωπαίων οι Δυτικοαφρικανοί έχουν δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να επιβιώσουν. Γερέρα, λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Αφρικανική Ήπειρος με ατυπικό χαρακτήρα χαρακτηρίζεται η Ήπειρος του πόνου αλλά σε αυτή την περίπτωση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτός ο χαρακτηρισμός με την έμπολα και τις γενοκτονίες ε, που ε, οδήγησαν στο να αποβιώσουν εκατομμύρια άτομα εκεί η φτώχεια, η ε, έλλειψη νερού υποδομών, η θνησιμότητα των παιδιών πλήττουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα σε αυτή την Ήπειρο υπάρχει και ένοπλη βία, υπάρχει τρομοκρατία υπάρχουν εμφύλοι πόλεμοι παντού Μία Ήπειρος που πριν από, δεκα, ε, πριν από κάποιες ε, δεκαετίες ε, κατάφερε να ξεφύγει από την κατάσταση της απικιοκρατίας, τώρα όμως βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Για αυτή την Ήπειρο τώρα, σε αυτή την Ήπειρο παρουσιάστηκε η μάστιγα του ιού της έμπολα. Και όπως ανέφερε η Επίτροπος η κυρία Γεωργίευα, έχει τρία χαρακτηριστικά αυτή η κατάσταση. Μία γεωμετρική αύξηση σε σχέση με τους όσους μολύνονται, υψηλότατο ποσοστό θνησιμότητας 60% και από την άλλη πλευρά απουσία υποδομών και δυνατοτήτων περίθαλψης με τις οποίες δυνατότητες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτές οι χώρες και αυτή είναι η πρόκληση να προσφέρουμε υποδομές να προσφέρουμε ιατρικό φαρμακευτικό υλικό και να επιτραπεί να υπάρξει δυνατότητα να δημιουργηθούν υποδομές να υποστηρίξουμε λοιπόν το Συμβούλιο του Μιλάνου να υποστηρίξουμε τις δράσεις των Ηνωμένων και τέλος να υποστηρίξουμε στις 24 Σεπτεμβρίου την απόφαση των χορηγών ώστε να διασφαλιστούν τα κονδύλια για αυτή τη δράση. Δύο τελευταία λόγια. Όσο το δυνατόν γοργότερα επικυρώσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης οι Ευρωπαίοι, τόσα περισσότερα κονδύλια θα έχουμε ώστε από πλευρά δομών και διαθρώσεων να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Φόρντ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα φέτος το κοινοβούλιο ε, μίλησε και μίλησα και εγώ για κλινικές δοκιμές όπου μιλάμε για τα 600 εκατομμύρια τα οποία ε, δαπανούμε κάθε χρόνο για να βρούμε κάποιες θεραπείες για επιδημίες οι οποίες θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν στην πηγή και που δημιουργούν όλο και μεγαλύτερους κινδύνους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό ε, να επιταχύνει την χρήση αυτών των κονδυλίων για κάποια εμβόλια, για παράδειγμα κατά του έμπολα ε, κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Κανεί δεν μπορεί να καταπολεμήσει τον έμπολα μόνο. Θα μπορέσουν λοιπόν έτσι οι Αφρικανοί ε, ε, φίλοι μα να συνεργαστούν με και ιδιωτικέ επιχειρήσει Γκλάξο Σμιθ για παράδειγμα, ή και με ευρωπαϊκού ερευνητέ, Ευρωπαίου με συγχωρείτε ερευνητέ, για να δούνε ποιο θα είναι το πιο, η πιο σύντομη δυνατότητα να αποκτήσουμε το εμβόλιο κατά του έμπολα. Έχουμε εμπειρογνώμονε που μα λένε πω ο έμπολα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ιό και πρέπει να σας πω πως έχουμε ήδη εξετάσει εμείς στην Επιτροπή μας τις ηθικές διαστάσεις αυτού του θέματος. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα και να καταφέρουμε να τα χρησιμοποιήσουν οι εμπειρογνώμονες όπως χρειάζεται ήδη. Σας έχουν σηκώσει δύο κάρτες. Ο κύριος Κάρβερ και η κυρία Μόη. Ε, θα απαντήσετε. Yes, okay. Ε, Ωραία. Κύριε Κάρβερ, πρώτος εσείς. Ευχαριστώ πολύ ε, που δέχεστε καταρχήν την ερώτησή μου. Θα ήθελα να πει, συνάδελφος, αν δέχεται τις απόψεις ε, τον όσων είπε ο κύριος Ντέβα που μίλησε για την κατανάλωση κρέματο, κρέατος από θυράματα που φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να μας πει τι κάνει το δικό της κόμμα γιατί νομίζω ήταν η δική της κυβέρνηση η οποία ε, ε, πρότεινε ε, να συγχωνευτούν κάποιες τελωνιακές υπηρεσίες οι οποίες πλέον δεν είναι οι υπηρεσίες φύλαξης της μεθορίου αλλά όπως λέμε χαρακτηριστικά στην Αγγλία της ε, μη φύλαξης της ε, μεθορίου. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν τι συμβαίνει. Εσείς από τις ε, υπηρεσίες τελωνίων αφαιρέσατε προσωπικό, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούν να ψάξουν καλά όσους γυρνούν από την Αφρική και ενδεχομένως έχουν μαζί τους αυτό το κρέας από θυράματα. Οι συνάδελφοί μου είπανε ότι αυτά τα λεφτά θα πρέπει να πάνε σε ερευνητές. Υπάρχει ένα σύστημα για να ελέγξουμε το πώς χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές αυτά τα λεφτά. Φερρυπίν στην ε, Ιταλία υπάρχει μεγάλη διαφθορά και σε αυτόν τον τομέα. Και οι ερευνητές συχνά ε, είναι στην τσέπη διαφόρων ε, παραγόντων των πανεπιστημίων και θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχουμε τα λεφτά που τους δίνουμε, ούτως ώστε να είμαστε και αποτελεσματικοί και να, αποτελεσ... να υπάρχουν και απτά αποτελέσματα. Φόρντ, έχετε το λόγο. Για την πρώτη ερώτηση να σας πω πως η αρχή που ακολουθούμε στο Κοινοβούλιο είναι ότι αν θέλεις να κάνεις ερώτηση σε άλλο μέλος του Κοινοβουλίου, το απευθύνει σε εκείνο το μέλος του Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να απαντήσω μια ερώτηση η οποία ουσιαστικά απευθύνεται στον κύριο Ντέβα. Γιατί πραγματικά είναι ένας αξιόλογος συνάδελφος, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω. Θα απαντήσω παρόλα αυτά θα απαντήσω παρόλα αυτά για το θέμα ε, του βρετανικού ρόλου ε, στο πρόγραμμα, στα ερευνητικά προγράμματα τα οποία μόλις περιέγραψα και για να απαντήσω στη δεύτερη αυτή ερώτηση τι να σας πω για τους Ιταλούς ερευνητές δεν έχω κάτι να πω η κοινότητα της Ευρωπαϊκής ε, με συγχωρείτε, η Βρετανική κοινότητα η ερευνητική είναι πραγματικά στην αιχμή του δόρετος προσπαθώντας να βρει λύσεις για τέτοιου είδους ε, μολυσματικές ασθένειες οι οποίες ε, δημιουργούν όλο και περισσότερους κινδύνους για τις δικές μας κοινότητες της χώρας μας. Για παράδειγμα, για τη φυματίωση η οποία είναι ανθεκτική στα ε, αντιβιωτικά, η οποία και πάλι κυκλοφορεί ανάμεσά μας και γι' αυτό οι δικοί μας ερευνητές ε, και οι εθνικές μας κυβερνήσεις ε, στοχεύουν στο να καλύψουν τις ασθένειες αυτές. Και πρέπει να σας πω πως το πρόγραμμά μας ε, δεν συμμετέχουν όλες οι εθνικές κυβερνήσεις, είναι ανοιχτό σε παραπάνω από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνεισφέρουν όλες αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε αυτά τα κονδύλια και να τα απευθύνουμε εκεί που χρειάζεται. Για δύο λεπτά η κυρία Σε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, το είπαν οι συνάδελφοι, θα το επαναλάβω κι εγώ. Βεβαίω χρειάζεται κινητοποίηση, διεθνή κινητοποίηση, επίγουσα κινητοποίηση κατά αυτή τη φρικτή πληγή και των επιπτώσεων που έχουν ήδη περιγραφεί οικονομικών, υγειονομικών, κοινωνικών αύριο. Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε, όταν θα τελειώσει η κρίση, γιατί είχαμε μια τόσο αργή απόκριση από την πλευρά της διεθνής, της κοινότητας. Πού βρε, ποια ήταν η δυσλειτουργία που δεν μας επέτρεψε να λάβουμε μια γρήγορη απόφαση και να έχουμε μια γρήγορη αντίδραση. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να χαιρετήσω τη δέσμευση του Προέδρου Ομπάμα. Χρειαζόμαστε μια στεναρή φωνή που να ασχοληθεί με το θέμα. Ξέρω τι κάνετε κύριε Επίτροπε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε στεναρή φωνή από πλευρά μας δεν ξέρω αν θα πρέπει να το Συμβούλιο ή η Επιτροπή, μια στεναρή φωνή που εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρώπη θα λάβει το λόγο για να μιλήσει για το τι πρέπει να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε τον έμπολα. Δεν έχει συμβεί και θα έπρεπε να γίνει. Τρίτο, εμεί συνεισφέρουμε χρηματικά θαυμάσια, αλλά δεν χρειαζόμαστε μόνο χρήματα επί τόπου. Όταν μιλάμε με το ιατρικό προσωπικό ε, και το υγειονομικό προσωπικό, μας λένε πως δεν μπορούν πια να ανταποκριθούν. Δεν είναι πολύ άριθμοι και χρειάζονται πιο συγκεκριμένη ε, βοήθεια, χρειάζονται προσωπικό, χρειάζονται εξοπλισμό, χρειάζονται κινητά εργαστήρια, χρειάζονται φάρμακα, χρειάζονται αεροδιακομιδές ακόμα και για τους ίδιους. Θα πρέπει εμείς λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβουμε αυτή τη μάχη και Τέλος, τέταρτη παρατήρηση, δεν θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει στις όμορες ε, και στις όμορες ε, χώρες για να κινητοποιηθούμε. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, για παράδειγμα, με το Μαλί, με το Κότ Τιβουάρ και να δούμε αν μπορούμε εκεί να ε, κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Και γι' αυτό πιστεύω πως η Ευρώπη θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ένα, ένα λεφτουδάκι η κυρία Μαρίνα. Μαλτιντού. Γινέα Κονάκρη, Σιέρα Λεόν, Λιβερία, χώρες που πλήττονται από επιδημία έμπολα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το οποίο καταστρέφει χιλιάδες ζωές. Θα πρέπει στον έμπορα να προσθέσουμε τη φτώχεια, γιατί υποφέρουν επειδή είναι χώρες φτωχές, ε, χώρες οι οποίες έχουν χάσει ε, τη θέση του στον κόσμο και πρέπει να σας πω πως για χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε γυρίσει την πλάτη της επιδημίας του έμπολα στην Αφρική και μόνο όταν είδε ότι μπορεί να φτάσει ακτέ μα μας ε, ο ιός και όταν τα τείχη μας και ε, οι προσπάθειες που έχουμε κάνει να κρατήσουμε την Αφρική εκτός τυχόν θα ε, κινδυνεύσουν, ε, έστρεψε το βλέμμα της προς την Αφρική. Φαίνεται πως δεν έχουν όλες οι ανθρώπινες ζωές την ίδια αξία. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν ασχολούνται με τις ασθένειες των φτωχών. Γιατί, Γιατί δεν είναι κερδοφόρες. Άρα λοιπόν οι οικονομικές ελίτ ε, ακολουθεί μια πολιτική εξίσου ε, θανατερεί με τα αποτελέσματα του έμπολα. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να συγχαρούμε την Κούβα που θα στείλει ιατρικό προσωπικό. Είναι η πιο μαζική αποστολή προσωπικού κατά του έμπολα. 165 άτομα, νοσοκόμες και γιατροί. Δείχνει για μια φορά ακόμα η Κούβα πως σε διεθνέ επίπεδο είναι η μόνη που προσφέρει αλληλεγγύη. Χέμπουκ, ε, για 1,5 λεπτό. Sehr verehrter Präsident, herzlichen Dank. Ich möchte noch einmal Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μία έκκληση. Ακούσαμε πάρα πολλά για τον έμπολα, για τις επιπτώσεις του, για την ανάγκη να βοηθήσουμε αυτές τις ε, χώρες, γιατί οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, ε, καθώς και οι κυβερνήσεις, ε, αισθάνονται ανήμπορες από το μέγεθος του προβλήματος. Δεν είναι θέμα αλληλεγγύης μόνο είναι κάτι πολύ παραπάνω, κάτι πολύ πέραν αυτού. Είναι καθήκον μας να διαθέσουμε ό,τι έχουμε στις χώρες αυτές. Το είπε κάποιος συνάδελφος. Έχουμε στρατιωτικό εξοπλισμό. Έχουμε στρατιωτικό προσωπικό επίσης, το οποίο μπορούμε να δώσουμε στα, στον ΟΗΕ για να βοηθήσουν αυτές τις χώρες προσωπικό το οποίο μπορεί να δουλέψει γιατί έχει κατάρτιση, έχει σοβαρή ιεραρχία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κι άλλο αν θέλουμε να περιορίσουμε αυτή την φοβερή καταστροφή ανθρωπιστική και άλλη. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν δράση δεν υπάρχει πια χώρος για, και χρόνος για συζητήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά τις συνέπειες εάν δεν περιορίσουμε τον έμπολα. Δεν θα είναι πια μόνο πρόβλημα υγείας. Δεν θέλω να επαναλάβω τα επιχειρήματα που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα. Σας παροτρύνω. Σας παρακαλώ να δράσετε τώρα. Για να δείξουμε σε όλους ότι δεν τους έχουμε απλώς το μυαλό μας και τη σκέψη μας, αλλά κάνουμε και κάτι γι' αυτό. Μελίν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η σοβαρότητα αυτής της επιδημίας του έμπολα θα πρέπει να προκαλέσει αυτόν τον προβληματισμό που πρέπει να κάνουμε για τον κίνδυνο πανδημιών στην Ευρώπη. Ξέρετε πως πάρα πολλά δεν έλαβε υπόψη η Ευρώπη. Ξέρετε πως εδώ και 50 χρόνια έχουμε τεράστια προβλήματα στη Μαύρη Αφρική με την διαφθορά, με την έλλειψη δομών υγείας και είδατε ότι καθυστερήσαμε και τρεις μήνες να διαγνώσουμε την επιδημία. Υπάρχουν κάποιες ε, ενισορροπίες μεταξύ Νότου και Βορρά. Έχουμε τις τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμών από Βορρά προς Νότο, χωρίς κανένα έλεγχο. Ξέρετε τι γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι επιδημίες να οδηγήσουν την Ευρώπη στο να αναλάβει τι ευθύνες γιατί μία πανδημία μπορεί να προβλεφτεί δεν είναι αναπόφευκτη. Είναι θέμα χρόνου. Θα πρέπει λοιπόν εκτός από τα μέτρα που λαμβάνουμε, πάντα έξι μήνες καθυστερημένοι εμείς εδώ στην Ολομέλεια, να αποφασίσουμε πως επιτέλους θα λάβουμε δράση. Πραγματική υγειονομική συνεργασία με τις χώρες που ε, είναι ε, σε τροχιά ανάπτυξη με τι αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να έχουν και τα δικά του συστήματα κοινωνικής προστασίας. Η μεταναστική πολιτική της Ευρώπης θα πρέπει να αναθεωρηθεί με υγειονομικού ελέγχου στα, στα σύνορα της Ευρώπης, αλλά και με συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με κέντρα υποδοχής υπό συνθήκες ιατρικής καραντίνας. Νομίζω ότι αυτό λένε και οι μεγάλοι επιδημιολόγοι της Ευρώπης και θα πρέπει επιτέλους να έχουμε ένα μεγάλο σχέδιο για να δημιουργήσουμε στην Ευρώπη την ίδια συγκεκριμένες ε, δομές για τέτοιου είδους ασθένειες με επιδημιολόγους γιατί καταλαβαίνετε πως ε, δεν θα ε, πρέπει να φτάσει το αύριο και να πει η Ευρώπη ότι δεν ανέλαβε τις ευθύνες της έναντι του, ενώπιον του τρίτου κόσμου. Σας παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο που έχετε. Γιατί αλλιώς θα καθυστερήσει η επόμενη συζήτηση. Δεν γίνεται έτσι. Ο κύριος Πίτερ Λίσε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ο ίδιος επί ένα χρονικό διάστημα εργαζόμουν ως ιατρό σε μια υποανάπτυξη χώρα. Γι' αυτό μπορώ να φανταστώ ακριβώς πώς αισθάνονται οι συνάδελφοι οι οποίοι αγωνίζονται σήμερα κατά του έμπολα, του ιού της έμπολα και έχουν ασθενείς και έχω κάθε σεβασμό για όλους που βοηθούν επί τόπου είναι πραγματικά έσχος ότι κάποιοι συνάδελφοι εδώ στο σώμα αυτή τη δύσκολη κατάσταση προσπαθούν κομματικά να την εκμεταλλευτούν. Τα ακούσαμε αυτά και τα θεωρώ απαράδεκτα δεδομένων των αναγκών και της ε, ένδυας των ανθρώπων σήμερα σε σχέση με τον ιό έμπολα. Δεν συμβαίνει το ότι οι άνθρωποι στην Ευρώπη <clears throat> πρέπει να φοβούνται όλοι ότι οι ίδιοι θα μολυνθούν ενδεχόμενα. Είναι καλό να δεχόμαστε ανθρώπους που βοήθησαν επί τόπου εκεί και να δοθεί η ασφάλεια ότι θα μπορέσουν να καλυφθούν οι ιατρικές τους ανάγκες με καλό τρόπο, με θετικό τρόπο και μπορούν σε σχέση με το καταδύναμη να θεωρούν οι πολίτες ότι είναι ασφαλείς. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μόνο επιταγή ανθρωπιστικής βοήθειας να βοηθήσουμε τους Δυτικοαφρικανούς αλλά κυρίως είναι μακροπρόθεσμα και προς το ίδιο το δικό μας συμφέρον. Διότι εδώ πολλές χώρες ε, βρίσκονται πρώτης κατάρρευσης. Ε. Δραματική είναι η κατάσταση σε αυτές τις χώρες και έχουμε πολλές κρίσεις παγκόσμια και γι' αυτό είναι προς το συμφέρον μας να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες ώστε να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους και να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να βοηθήσουμε. Είναι καλό ότι η Επιτροπή, κυρία Επίτροπε και πολλοί άλλοι ότι βοήθησαν να αυξηθούν τα κονδύλια Όμω θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο, ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα με τον προπολογισμό μα με αυτή την κατάσταση. Τις τελευταίες ημέρες επανειλημμένα άκουσα από τα κράτη-μέλη και από την χώρα από την οποία προέρχομαι ότι πρέπει να κάνουμε λέει, περισσότερα για την Ουκρανία, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για το Ιράκ, αλλά πρέπει να κάνουμε και περισσότερα και για την Δυτική Αφρική. Ο Τζοβάνι Λαβία, ο Ράιμε Μπέργκερ και όλοι όσοι ήταν εδώ και μάλιστα σε σχέση με τα όσα δεν προβλεπόντουσαν πρέπει να συζητήσουμε, να είναι πιο ευέλικτο το Συμβούλιο ώστε να μπορούμε αποτελεσματικά να αντιδρούμε σε τέτοιες κρίσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή. 1,5 λεπτό αρένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι έξαλλη, όχι για το θέμα της Κούβας, αλλά για το θέμα ε, της χειραγώγησης που γίνεται για τον έμπολα για να μιλήσει ο κόσμος για την μετανάστευση. Από το Μάρτιο οι γιατροί χωρίς σύνορα, χωρίς μας μιλάνε για τον κίνο του ιού και της επιδημίας. Έχουμε φτάσει τώρα το Σεπτέμβριο, έξι μήνες μετά. Και ο ιός εξαπλώνεται εκθετικά διπλασιάζεται ο αριθμός των μολυσμένων ανθρώπων κάθε 15 μέρες. Υπάρχει λοιπόν κατεπίγουσα ανάγκη να αντιδράσουμε. Ε, γιατί θα, το μετανιώσουμε να δρανήσουμε. Σήμερα θα πρέπει να διρωτηθούμε ως προς το τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να σταματήσει αυτή η ιστορία. Εγώ θα έλεγα απλά τα πράγματα. Οι γιατροί χωρίς σύνορα μας είπαν πολύ συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε μία συντονισμένη προσέγγιση, πρέπει να δώσουμε εξοπλισμό, χρειαζόμαστε καραντίνες, χρειαζόμαστε νοσοκομεία εκστρατείας, χρειαζόμαστε εργαστήρια, χρειαζόμαστε αερογέφυρες. Όλα αυτά τα κράτη-μέλη τα έχουν και ως σε επίπεδο αστικό αλλά και σε επίπεδο στρατιωτικό. Όταν μιλάμε για το στρατό, θα ήθελα να υπάρχουν και ανθρωπιστικοί στρατοί οι οποίοι υποστηρίζουν τους ε, χυμαζόμενους πληθυσμούς. Ας μην κλείνουμε τα αυτιά όλα τα μέσα είναι χρήσιμα για να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό, για να καταπολεμήσουμε αυτή την επιδημία. Ζητάμε από το Συμβούλιο αλλά και από την Κομισιόν να διαθέσουν αυτά τα μέσα στους πληθυσμού που χυμάζονται το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. per un minuto. Ευχαριστώ πολύ. Οι συνάδελφοί μου το έκαναν ήδη και δεδομένη σοβαρότητα τη κατάσταση δεν θα επανέλθω στα αριθμητικά στοιχεία τα οποία όλοι γνωρίζουμε και νομίζω ότι όλοι ε, δηλώνουν ότι έχουν υποεκτιμηθεί. Η καθυστερημένη απόκριση δική μα είναι αυτή η οποία με ανησυχεί. Νομίζω ότι όλοι το δέχονται αυτό, το είπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και εσείς κύριε Επίτροπε και ο κύριος Ομπάμα και αυτός ο δικός ε, χάρτης, η έρευνα και τα λοιπά, το σχέδιο δράσης θα χρειαστούν χρόνο. Εν τω μεταξύ λοιπόν η χώρα μας, για παράδειγμα ε, το Βέλγιο έχει την δυνατότητα να παρέμβει γρήγορα είτε στρατιωτικά είτε με πολιτικό προσωπικό για να αντιμετωπίσει αυτού ε, του είδους τις ανθρωπιστικές κρίσει. Όλοι οι επιτόπου μας λένε πως χρειάζεται συντονισμός και σε επιτόπιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ και πολύ καιρό μιλάμε για συντονισμό, το ξέρουμε, αλλά εκεί το είπε η κυρία Ριβάζη που έχει στείλει τα παιδιά της στην πρώτη γραμμή. Δεν βλέπουν συντονισμό από εμά και χρειάζονται κάτι παραπάνω και να δράσουμε πιο γρήγορα στην πραγματικότητα δεν έχουμε επιλογές κύριε Πρόεδρε. Αν θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε ο ιός αυτός να εξαπλωθεί και στην Αφρική και στις χώρες μας θα πρέπει και εμείς να δείξουμε αλληλεγγύη. Γιατί βέβαια αυτό δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά καθήκον. Η Φρανσουάς Γκροστέτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Βεβαίω αυτό το έχουν πει πολλοί συνάδελφοι πριν από μένα και βλέπουμε και ποιε είναι οι προοπτικέ και οι προβλέψει του ΠΟΕ για την εξάπλωση του έμπολα. Νομίζω είναι πολύ απεσιόδοξε. Α μην ξεχαστούμε. Δεν είναι μόνο πρόβλημα της Δυτικής Αφρικής. Ε, δεδομένου του μεγέθους αυτής της επιδημίας μας αφορά όλους. Έφτασε η στιγμή να κινητοποιηθούμε. Ε, την τελευταία στιγμή, γιατί χάσαμε ήδη πάρα πολύ θα ήταν τόσο εύκολο να αποποιηθούμε των ευθυνών μας και να πούμε η ασθένεια αυτή δεν επηρεάζει άμεσα ε, τη δική μας Ήπειρο. Μα ξέρετε πως είναι μια πραγματική παγκόσμια κρίση. Οι αξίες στις οποίες υπερασπιζόμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι στον κόσμο είναι η ελληνική, η αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμό αυτών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στηρίξουμε τις εμπλεκόμενες χώρες. Είναι μια υποχρέωση ηθική δική μας. Να υπογραμμίσω λοιπόν πως έχουν γίνει προσπάθειες από ε, το ιατρικό προσωπικό επιτόπου, από μη καπαόμικρον και είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε όσο μπορούμε. Να ξεπεράσουμε λοιπόν ε, την προστασία, όχι μόνο ε, το θέμα της προστασίας των αξιών που πρεσβεύουμε, αλλά και του ε, πληθυσμό μας, γιατί πραγματικά μιλάμε για μια ε, κρίση ε, χωρίς προηγούμενο. Υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης μιας ολόκληρης περιφέρειας, κοινωνικά, οικονομικά και ανθρωπιστικά. Η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραμείνει παθητικός εταίρος ε, ενώπιον ενός τέτοιου δράματος. Γιατί αυτό σημαίνει Ευρώπη για τους συμπολίτε μας. Μια Ευρώπη η οποία χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες που έχει παγκόσμιο επίπεδο και η οποία είναι υπεύθυνη για τη δράση. Ας αναρωτηθούμε. Ο ιός του έμπολα ανακαλύφθηκε το 76 και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε ερωτήματα. Θα πρέπει περισσότερο από ποτέ και κλείνω να προωθήσουμε την έρευνα ε, στο χώρο της ιατρικής. Είναι απαραίτητο καινοτομία, ιατρική πρόοδος, αλληλεγγύη ευρωπαϊκή, η επιδημία του έμπολα εκτός από σκέτη υγειονομική κρίση, είναι μια κρίση ε, η οποία χρειάζεται μια απόκριση από την ίδια την Ευρώπη. Ζιλ Πάνιο, 1,5 λεπτό. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, ναι, είναι κατεπήγον το θέμα. Το είπαν προηγούμενοι συνάδελφοι, 20.000 άτομα είναι πιθανά θύματα ή θα είναι πιθανά θύματα μέχρι το τέλος του 2014. Να μην το ξεχνάμε όμως, ένα εκατομμύριο Αφρικανοί είναι σε καραντίνα σήμερα λόγω της επιδημίας. Είναι κατεπήγον το πρόβλημα και χαίρομαι που η Κομισιόν απεμπλόκαρε 152 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά σήμερα πρέπει να μας πει πολύ συγκεκριμένα σε τι θα χρησιμεύσουν αυτά τα λεφτά. Καταρχάς πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των κέντρων θεραπείας ε, που έχουν στη διάθεσή τους ε, δυνατότητες ε, καραντίνας. Να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, κινητά εργαστήρια, αερογέφυρες, περιφερειακά περιφερειακά κέντρα θεραπείας. Αυτά μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Εγώ ήμουν ε, εισηγητής ε, της έκθεσης για τις ε, διασυνοριακές σοβαρές απειλές στην υγεία που υιοθετήσαμε τον Ιούλιο του 2013 και που ε, τέθηκε σε ισχύ 6 Νοεμβρίου του 2013. Και ως εισηγητής θεωρώ ότι ήγηκε η ώρα τα κράτη-μέλη να οργανώσουν πολύ γρήγορα μια έκτακτη συνεδρίαση των ε, Υπουργών Υγείας για να συζητήσουν για αυτή την πανδημία. Θα πρέπει, όπως λέει και η απόφαση για τις διασυνοριακές απειλές για την υγεία, ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε το συντομότερο δυνατό, δυνατόν να δούμε τι ε, οι ιατρικές εγκαταστάσεις υπάρχουν που μπορούν να υποδεχτούν ασθενείς, να ενεργοποιήσουν το δίκτυο το ευρωπαϊκό Εργαστήριο που μπορεί να ανοιχνεύσει τους παθογόνους οργανισμούς και να είμαστε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης των Ασθενειών. Αυτά είναι, κύριε Επίτροπε, τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν τώρα. Μπέρτερ, για ένα λεπτό διπλασιάζονται κάθε τρει εβδομάδες τα κρούσματα έμπολα. Ενδεχομένω λοιπόν θα έχουμε και εδώ κάποιε επίγουσες καταστάσεις, μια και ξεπερνά τα όρια. Ξεκινήσαμε να κινητοποιούμεθα, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα αποφύγουμε και ε, μελλοντικές τέτοιες επιδημίες. Χρειαζόμαστε θεραπείες όχι μόνο για τον έμπολα αλλά και για άλλες θανατηφόρες ασθένειες. Αυτές ε, τις ασθένειες δεν τις, ε, με αυτές τις ασθένειες δεν ασχολούνται φαρμακευτικές εταιρείες γιατί δεν υπάρχει κέρδος. Ξέρετε πως η ελονοσία και το εμβόλιο ε, για την ελονοσία αυτή τη στιγμή τρέχει από μια εταιρεία που οποία είναι έτοιμη να παρουσιάσει και κάτι αντίστοιχο για τον έμπολα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε μέσω των δικών μας ερευνητών και μέσω των δικών μας ερευνητικών κονδυλίων ε, τις προσπάθειες που γίνονται σε αυτό το χώρο για να περιορίζουμε αμέσως τις ε, επιδημίες και αυτό μέσω εκπαίδευσης χρησιμοποιούμε την πραγματογνωμοσύνη μας και εκπαιδεύουμε τους εμπειρογνώμους έτσι ώστε όταν θα ξανασηκώσει το κεφάλι της αυτή η επιδημία θα είμαστε έτοιμοι ε, να ε, την περιορίσουμε. 1,5 λεπτό λαβία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία ε, Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα καταρχήν να στρέψω μία σκέψη για τα χιλιάδες θύματα της επιδημίας. Και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα άτομα τα που είναι γιατροί, νοσοκόμοι, εθελοντές και συνεργάζονται για να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την αρρώστια και προς τον συμφέρον των δικών μας ευρωπαϊκών χωρών. Τώρα πρέπει να μιλήσω για τους πόρους που διαθέτουμε. Ξέρουμε ότι για να παρέμβουμε γρήγορα και για να έχουμε μια έντονη απάντηση χρειαζόμαστε πόρους. Οι πόροι κινητοποιούν ε, μέσα και άτομα ε, προς το συμφέρον των ε, πληθυσμών αυτών. Δυστυχώς Πόρου έχουμε λίγους πια στην Ευρώπη. Γιατί, Γιατί στο πολιτεύσιμο-συνομικό πλαίσιο δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια ευελιξίας. Αυτό θα πρέπει να μα οθήσει στη διαπραγμάτευση του προπολογισμού που κάνουμε να δούμε ποιοι είναι οι απαραίτητοι πόροι ε, και να, να τους πάρουμε και από, αν χρειαστεί, και από κάποια προγράμματα που δεν είναι τόσο απαραίτητα. Επιτρέψτε μου ως ε, πρόεδρος της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, Υγείας στο Συμβούλιο Υπουργών στο Μιλάνο τη Δευτέρα να κάνουμε μια έκτακτη προσπάθεια και 28 χώρες ούτω ώστε να υπάρξει μια συντονισμένη παρέμβαση, άμεση παρέμβαση για μια τέτοια επιδημία όπως αυτή. Σήμερα δεν μας αφορά άμεσα, αλλά σίγουρα πρέπει να παρέμβουμε χωρίς να χάσουμε χρόνο για να μπορέσουμε να προλάβουμε τα προβλήματα τα οποία θα έχουμε εάν δεν κάνουμε τίποτα και στην Υπηρώ μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Φαν Μπρέμπτε, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εγώ σε αυτό το σύντομο διάστημα που έχω για την παρέμβασή μου ένα μόνο σημείο θα αναφέρω που αναφέρθηκε και από συναδέλφου, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ο συντονισμό είναι αυτό το σημείο μεταξύ των προσπαθειών μας και στον κύριο συντονιστή. Τον κύριο συντονιστή των Ηνωμένων Εθνών θέλω να αναφέρω. Παράθεμα είπε ο συντονισμό σώζει ανθρώπινε ζωέ και ο συντονισμό φυσικά αφορά και την ιατρική παρακολούθηση, ε, όλη την επιμελητιακή υποστήριξη και βοήθεια, την τροφοδοσία, όλη αυτή την προστασία που είναι αναγκαία και πρέπει να παρασχεθεί. Για τους υπεύθυνους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη πραγματικά παρακάλεσαν, παρακλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην δρουν μεμονωμένα και ξεχωριστά, αλλά ενωμένα και με συντονισμένο τρόπο. Άλλαξε κάτι. Η επιδημία άρχισε να παίρνει τώρα δραματικές διαστάσεις και στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Απαριθμίσατε ποιες πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν και ποιες δράσεις γίνονται. Με τις καλύτερες προθέσεις το κάνατε αυτό, σίγουρα. Αλλά στο μέλλον ταχύτερα, πολύ ταχύτερα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συντονιστικός φορέας να δράσει και να μεριμνά ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι σημαντικό και για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό. Να συμμετέχει η Ευρώπη με ισχυρό τρόπο, με συντονισμένο τρόπο ώστε να είμαστε ισχυροί στην παγκόσμια σκηνή, ώστε η πραγματογνωμοσύνη να μπορεί να συντονίζεται και να είναι αποτελεσματική, ώστε μια ανθρωπιστική βοήθεια να παρέχεται και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή αυτή τη Αφρική. Ευχαριστώ. Ε, Μπεθερίλ. λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να ξεκινήσω στηρίζοντας ε, τα θύματα του έμπολα και να πω πως θα στηρίξουμε επίσης και όσους εργάζονται επί τόπου διακινδυνεύοντας τη ζωή τους για να σώσουν α, ζωές ανθρώπων που ζουν σε χώρες που δεν έχουν καν τις ελάχιστες υποδομές για να ξεπεράσουν αυτή την ε, ε, επιδημία. Ο Μιγγέλ Πάχαρες, ένας Ισπανός παπάς, έχασε τη ζωή του μολυσμένος στη Λιβερία βοηθώντας τους ε, ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Και ξέρεις πως αυτοί οι, αυτά τα άτομα τα διώχνουν οι ίδιες τους οι κοινότητες επειδή φοβούνται ότι θα μολυνθούν. Δεν υπάρχει δημόσια υγεία στις χώρες αυτές. Χρειάζεται μια διεθνή συντονισμένη απόκριση και θα πρέπει να εργαστούμε πιο γρήγορα γιατί 2.500 ζωές έχουν ήδη χαθεί με στη σιωπή και η κατάσταση χειροτερεύει καθημερινά. Ο ιός του έμπολα έχει καταστρέψει τις αδύναμες ήδη οικονομίες έχουν η συνέχεια αυξανόμενε ανθρωπιστικέ ανάγκε, οικονομικέ ανάγκε, και τα πράγματα θα χειροτερεύσουν. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε αυτή την ασθένεια. Ο αριθμό των ασθενών ε, αυξάνεται πιο γρήγορα από τη δική μα δυνατότητα να βοηθήσουμε. Χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά θα πρέπει να στείλουμε και περισσότερους εμπειρογνώμονε στην περιοχή. Θα πρέπει όλε οι χώρε να ασχοληθούν με το θέμα τη έρευνα και να μην ξεχάσουμε και τα μέτρα που θα περιορίσουν την εξάπλωση τη επιδημία. Δεν θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να καταδικάσουμε τις χώρες αυτές οι οποίες ήδη έχουν χάσει κάθε ελπίδα να βγουν από τη φτώχεια, να μην τις απομονώσουμε και θα κλείσω υπενθυμίζοντάς σας πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν αυτούς τους ασθενείς. Τα άτομα αυτά χρειάζεται ε, να αναγνωριστούν από εμάς ανεξάρτητα με το αν είναι Ευρωπαίοι, Αμερικανοί ή Αφρικανοί. Είναι οι ήρωες οι δικοί μας, οι ανώνυμοι ήρωες και σε αυτούς εμείς θα πρέπει όχι μόνο να αφιερώσουμε την προσοχή μας αλλά και την ε, πολύ γρήγορη δράση που πρέπει σύντομα να αναλάβουμε. Κυρία Σάντεμος, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η επιδημία της έμπολα είναι μια παγκόσμια πρόκληση και γι' αυτό είναι πολύ καλό να διασφαλίσουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη τώρα επιτέλους ε, ξεκινούν να αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα αυτό το πρόβλημα και να δραστηριοποιούνται. Επιτέλους ήθε, ήταν η χρονική στιγμή να γίνει αυτό. Δύο εκκλήσεις, μία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία προς τα κράτη-μέλη. Πρώτον, το πρόβλημα της εκένωσης ε, του ιατρικού προσωπικού Πρέπει να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Είναι η μόνη δυνατότητα που υπάρχει ώστε να μπορέσουν να αποσταλούν περισσότεροι από πλευρά ιατρικού προσωπικού να τους αντικαταστήσουν. Και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τα κονδύλια, τα χρήματα εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν δεν θα αντληθούν από την κλασική βοήθεια για την ανάπτυξη και τα κονδύλια για την αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει να είναι νοπό χρήμα. Διαφορετικά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη αυτά ώστε μακροπρόθεσμα να ανοικοδομήσουν το ιατρικό του σύστημα και τι υποδομέ του. Χρειάζεται μαζική βοήθεια, αλλά πρέπει με το σωστό τρόπο να δράσουμε. Ελπίζω ότι σωστά θα μπορέσουμε να συντονιστούμε ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια Σράγερ πήρε και 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πράγματι έχουμε δει ε, χιλιάδες από το πρόβλημα αυτό στην Αφρική και δυστυχώς χιλιάδες ανθρώπων κινδυνεύουν να αμολυνθούν. Αυτές οι χώρες ήδη υποφέρουν, οι οικονομίες τους έχουν φυγεί σοβαρότατα και διαρωτώ με τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς στην Ευρώπη για να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν συζητήσεις και ο Υπουργός Υγείας είπε ότι απαιτούνται αγορές μαζικές εμβολίων. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλος του προβλήματος γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην κυκλοφορία ενός εμβολίου. Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις έρευνες αυτές. Είναι εξίσου σημαντικό το θέμα με το πρόβλημα του έμπολα αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Μίτσι, ένα λεπτό. Ήδη από την αρχή του χρόνου ο ιός εμπόλα έχει προκαλέσει 2.500 νεκρούς και στη Λιβερία και στη Σιέρα Λεόν, αλλά έχουν φυγεί και η Νιγηρία και από ό,τι φαίνεται η Σενεγάλη. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση ε, του ιού αυτού, αλλά δυστυχώς η διεθνής ανταπόκριση είναι ανεπαρκής. Το πρόβλημα αφορά τις ζωές των συνανθρώπων μας. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Έχουμε καθήκον απέναντι στα θύματα και στις οικογένειές τους και φυσικά και ανάμεσα στους επαγγελματίες της υγείας που τους φροντίζουν να πάρουμε μέτρα. Απευθύνω έκκληση λοιπόν στην Ιταλική Προεδρία όπως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουν κάθε προτεραιότητα στην καταπολέμηση αυτής της μάστιγας και να οργανώσουν το ταχύτερο δυνατόν ε, μια συνάντηση κορυφής που να ασχοληθεί με το θέμα. Απαιτούνται μέτρα για να περιοριστεί η επιδημία. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να πεθάνουν περισσότεροι ώσπου να δράσουμε. Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Να εκριζωθεί η απειλή αυτή από την Αφρικανική Ήπειρο και να διαβεβαιώσουμε τους πληθυσμούς ότι θα τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε λέει, ναι, κυρία Κιέγκε. Καμία χώρα δεν θα πρέπει να αφαιθεί ε, μόνη. Τέτοιες ασθένειες μπορούν να αντιμετωπιστούν, αλλά αυτό απαιτεί συγκεκριμένη και συντονισμένη δράση σε διεθνές επίπεδο. Ο περιορισμός απλά της ασθένειας δεν είναι μια επιλογή σωστή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες της ασθένειας και να ενισχύσουμε τα συστήματα υγείας των χωρών αυτών τα οποία είναι ανεπαρκέστατα. Είναι κάτι το οποίο θα θέσει σε απειλή την ανάπτυξη αυτού του τμήματος της Αφρικανικής ε, Ήπειρου. Τέτοιες τραγωδίες στο μέλλον θα πρέπει να αποφευχθούν. Εδώ έρχεται φυσικά η καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία είναι ε, πάρα πολύ σημαντική θα πρέπει να βοηθήσουμε την κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού επιτόπου, να βοηθήσουμε στην κατασκευή, στην οικοδόμηση νέων εγκαταστάσεων και είναι απαράδεκτο ε, μια χώρα σαν την Λιβερία να θέτει σε καραντίνα ένα ολόκληρο τμήμα της πρωτεύουσας της χώρας. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Ο κόσμος σας είναι παγκοσμιοποιημένος και θα πρέπει να αναλάβουμε δράση άμεσα. Περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye. Ένα λεπτό, όχι περισσότερο. Μίκολα Σικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, το θέμα αυτό της έμπολα συγκρίνεται μόνο με τη... την πανούκλα στο Μεσαίωνα. Έτσι, οι χώρες, η Λιβερία συγκεκριμένα είναι πάντα στα όρια της κατάρρευσης μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και εμείς οι γιατροί μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει εμβόλιο ή φάρμακο. Το ψάχνουμε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασχοληθεί λίγο πιο σοβαρά με το θέμα και να βρει μια λύση. Όχι μόνο στο προληπτικό τομέα ή μέσω επιδημιολογικών μέτρων, αλλά να δείξουμε και περισσότερη αλληλεγγύη. Είναι και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι και υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει των πλησίον στην Αφρική ebola a provocat decesul a aproape trei de persoane iar alte cel puțin două de persoane. Ο κύριος Γκρέσκο, κοιτάξτε, η έμπολα προκαλεί χιλιάδες θανάτους στην Αφρική, αλλά το θέμα είναι σοβαρό. Δηλαδή, εμείς ακούμε χιλιάδες ανθρώπους, αλλά είναι άνθρωποι, δεν είναι αριθμοί. Θα ήθελα επίσης ε, βεβαίως ε, και εγώ να πω πως πρέπει να ενισχύσουμε ιδιαίτερα για τον ιό και να συνεργαστούμε με τους διεθνείς μας εταίρους και να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κάτι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει το πρόβλημα. Όπως μας λένε οι εταίροι μας στη Δυτική Αφρική, δεν υπάρχει δυνατότητα να διαχειριστούμε την ασθένεια, να διαχειριστούν την ασθένεια εκεί καλύτερα. Αν σκεφτούμε δε ότι έχουν περικοπεί και τα κονδύλια τα αναπτυξιακά της Ένωσης, τι να κάνουνε. Πρέπει να αντιδράσουμε. Καλές οι δεσμεύσεις του Κομισιόν, αλλά πρέπει να στείλουμε και κάνα φράγκο εκεί πέρα. έχουμε αφήσει μόνο τους γιατρούς χωρίς σύνορα και κάτι τέτοιους ανθρωπιστικούς οργανισμούς. Αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις επιδημίες αυτές έχουν ανάγκη από τη βοήθειά μας. Η επιδημία αυτή είναι μια τρομακτική απειλή για την υγεία στο σύνολο της περιοχής και όχι σε συγκεκριμένες χώρες. Η αλήθεια είναι ότι οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι οι οποίοι τροφοδοτήθηκαν από το καπιταλιστικό και στρατιωτικό status quo οδήγησαν σε πολιτικές λιτότητας οι οποίες επιδεινώνουν την κατάσταση. Χώρες όπως η Σιέρα Λεόνε, η Λιβερία, η Γουινέα, η Νιγερία είναι χώρες οι οποίες υπέστησαν τον ζυγό της απεικιοκρατίας και αμέσως μετά τον ζυγό του υπεριαλισμού. Ε, αυτό τις οδήγησε στην καταστροφή. Πρόκειται για χώρες οι οποίες δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την επιδημία αυτή σήμερα. Έχουν λοιπόν την υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε λόγω των χρεών του παρελθόντος να αναλάβουν αποτελεσματική δράση. Θέλω να σημειωθεί εδώ η διαφορά ανάμεσα στη ΣΥΠΑ που στέλνει στρατιωτικό προσωπικό και στην Κούβα που στέλνει αυστηρά ιατρικό προσωπικό στις περιοχές αυτές. Äh, Κύριε Πρόεδρε, είχαμε μία ακρόαση με τον αρμόδιο επίτροπο και απαιτήσαμε περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα. Είναι λυπηρό, ειδικά όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση τέτοιων εκτάκτων περιπτώσεων, ε, να είναι τόσο συγκρατημένα τα κρατημέλη. Τέλο πάντων, κάλλιο αργά παρά ποτέ πρέπει να πούμε στο Συμβούλιο, αλλά στο μέλλον δεν πρέπει να επαναληφθούν αυτέ οι καταστάσει Τώρα, αυτά τα λαϊκίστικα που ακούγονται δεν βοηθάνε καθόλου εκεί κάτω στην Αφρική. Πρέπει να, έχουμε, να ξέρουμε πώς θα εκδηλώνονται συχνότερα αυτές οι επιδημίες και αντί να θρηνεί η Ευρώπη καλά θα κάνει να ανασκουμποθεί και να βοηθήσει και βεβαίως έρευνα και ανάπτυξη, αυτό ακούστηκε από όλους, να δούμε τι θα κάνουμε. Etheridge. Ευχαριστώ. Καθώς παρακολουθούμε την τρομεκτική αυτή ιστορία και το πρόβλημα να γίνεται συνεχώς χειρότερο, μπορούμε όλοι μαζί να πούμε ότι χαιρετίζουμε όσους προσπαθούν εκεί να σώσουν τον άρρωστο κόσμο και τα παιδιά και οι πολιτικοί θα έπρεπε να προσπαθήσουν να βρουν τίμιες και ειλικρινείς, να κάνουν τίμιες και ειλικρινείς προτάσεις για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτό το φοβερό πρόβλημα. Πάνω απ' όλα θα έπρεπε ενωμένοι να στείλουμε ευχές και προσευχές και τις ελπίδες μας σε όλους όσοι υποφέρουν από αυτό το τρομερό πράγμα. Αυτό είναι το βασικό που μπορούσαμε να πούμε από εδώ σήμερα. κύριος Βόιτ. Όχι μόη, void. Α, καλά, με συγχωρείτε, κατάλαβα μόη. Ναι, κυρία Επίτροπε, έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για το τρίτο πράγμα που είπατε. Είπατε πως ο ιός πρέπει να απομονωθεί και να καταπολεμηθεί, αλλά ο ιός, όχι οι χώρες. Αλλά βεβαίως οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείε πετάνε σε αυτές τις χώρες. Ε, είναι υπεύθυνη συμπεριφορά αυτή θεωρείτε εσείς ή ανεύθυνη. Γιατί ο ιός δεν σταματάει. Άμα φτάσει κάποιος ε, φορέας ε, στο Βερολίνο, στο Παρίσι ή στις Βρυξέλλες, δεν θα μπορέσουμε να φροντίσουμε τις άλλες χώρες, θα έχουμε εμείς το πρόβλημα. Συγκεκριμένα λοιπόν ρωτάω, ψάχνουμε τους ανθρώπους, υπάρχει δυνατότητα τον προσγειώνονται τα αεροπλάνα και να υπάρχει μια απομόνωση, μια καραντίνα μέχρι να δούμε αν είναι ασθενής ή όχι. Γιατί αλλιώς η κατάσταση ενδείκνυται για λαϊκισμό. Γιατί άμα δεν δράσουμε εγκαίρως και φτάσει ο ιός στην Ευρώπη, είναι πάρα πολύ αργά. Τελεί. Ονορεύει Γιάκοβτσιτς. Γιάκοβτσιτς. Poštovane dame i gospodo, prije svega bih se htio zahvaliti Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω εκείνους που εργάζονται επί τόπου για, στις χώρες όπου έχει ξεσπάσει αυτή η πανδημία και προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωσή της. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η πανδημία αυτή μας εξέπληξε. και βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στο συντονισμό της αντιμετώπισης της. και εμείς όλοι μαζί αλλά και εταίροι μας εκτός Ένωσης πρέπει να συντονιστούμε γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη Δυτική Αφρική, στην Ευρώπη, ισχύει για ολόκληρο τον πλανήτη. Γι' αυτό είμαι υπέρ της ενίσχυσης της έρευνας και για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι τόσο δραματική η κατάσταση που μας λένε οι γιατροί πως χρειάζονται ε, στρατιώτες και μάλιστα διατεθειμένοι να πυροβολούν. Εντάξει και λεφτά, αλλά αν ε, στείλουμε εκεί πέρα ανθρώπους χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο θα κάνουμε χειρότερη την κατάσταση. Ο ΙΕ πρέπει εδώ πέρα να αναλάβει μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση κινητά νοσοκομεία, φάρμακα, γιατρούς και ειδικού και στρατιώτες οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να προστατεύουν αυτούς τους ανθρώπους γιατί έχουν υποστεί και επιθέσεις. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα λοιπόν πριν εξαπλωθεί η επιδημία. Για τερμά και έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο ιός αυτός στην παρούσα φάση είναι το μείζον πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η περιοχή. Οι διεθνείς οργανισμοί δεν έλαβαν σοβαρά όσο έπρεπε την απειλή αυτή και ο ιός κέρδισε έδαφος και κατέκτησε και νέες περιοχές. Σήμερα οι διεθνείς οργανώσεις θα πρέπει να συντονίσουν τις δράσεις τους. Είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένο γιατί βλέπω ότι ο ΠΟΕ δεν έχει επαρκείς πόρους στην διάθεσή του για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Θα ήθελα όμως σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διεθνές, διεθνείς συγγνώμη, οργανώσεις όπως ο να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια βήματα και να αποκτήσουμε τους κατάλληλους πόρους. Τελευταία παρουσίαση. θα θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας απέναντι σε όλες τις ε, οικογένειες οι οποίες υποφέρουν στις περιοχές αυτές από τον ιό αυτό. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, αποφασίσει να στείλουν 150 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος τα πήρε τα χρήματα αυτά, τι τα κάνανε μέχρι τώρα και τι θα γίνουν τα χρήματα αν στείλουμε μάλιστα και άλλα. Θα ήθελα λοιπόν παρακαλώ στην περίπτωση που αποσταλούν και στην Ιταλία τα χρήματα αυτά, θα ήθελα να μας πείτε πώς θα αποφύγετε να τύχουν να γίνουν λία της κομπίνας και της απάτης που επικρατεί στη χώρα μου. Η Επίτροπος Γεωργίδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έλαβαν το λόγο. Θα αρχίσω από το κατά πόσον η Ευρώπη αντέδρασε αρκετά γρήγορα. Από ανθρωπιστική πλευρά ναι, ναι. Ήμασταν οι πρώτοι που χορηγήσαμε χρηματοδοτική βοήθεια και στείλαμε προσωπικό και γιατρούς που ρισκάρουν τη ζωή τους εκεί επί τόπου ώστε να δοθεί προσοχή σε αυτή την επιδημία. Και από τον Μάρτιο που οπότε και άρχισε επανειλημμένως κάναμε ανθρωπιστικές παρεμβάσεις δηλώνοντας προς όλους ότι είναι σοβαρά τα πράγματα και ότι πρέπει να αντιδράσουμε με συντονισμένο τρόπο. Τον Αύγουστο, μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πλησιάσαμε τα κράτη-μέλη μέσω του μηχανισμού ε, πολιτικής προστασίας για να προστατευτούν συγκεκριμένες κοινότητες. Πολύ συχνά όμως είμαστε σαν την καλαμιά στον κάμπο μόνοι μας. Είμαστε μάλλον αυτοί που πρώτοι ως φωνή βόντος εν τη ερήμο προειδοποιούμε και δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα μπορεί να πει κανεί ότι δεν ανταποκριθήκαμε αρκετά γρήγορα συνολικά α, στις εκκλήσεις των γιατρών και ιδιαίτερα των γιατρών χωρίς σύνορα. Αλλά χρειάστηκε χρόνος για να αναγνωρίσει ο κόσμος. Ακόμη και ο ΠΟΗ, ο Υπαγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, χρειάστηκε χρόνο για να αναγνωρίσει πόσο σοβαρά είναι αυτά τα πράγματα να παραδεχτεί. Γι' αυτό θα ήθελα να επενέσω τα κράτη-μέλη, διότι τις τελευταίες εβδομάδες αντέδρασαν και αυτά. Η Αυστρία παραδειγματος χάρη έστειλε προστατευτικά μηχανήματα, η Ιταλία οργάνωση νοσοκομείων, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία νέα κέντρα, θα ανοίξουν νέα κέντρα περίθαλψης. Η Ουγγαρία βοήθεια σε είδο Η Ισπανία στη Σιέρα Λεόν παρενεύει και λοιπά και λοιπά και επίσης έχουμε και τους στρατιωτικούς μας που ερευνούν πώς να βοηθήσουν στην εκένωση πληθυσμών που το χρειάζονται. Το είπατε και εσείς πολλές φορές. Έτσι λοιπόν τελικά βλέπουμε ότι γενικά αρχίζει, υπάρχει κινητοποίηση. Αλλά πρέπει να διατηρήσουμε την προσοχή αυτή στο θέμα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κρίσεις παράλληλες και πολύπλευρες και μπορεί να τεθεί θέμα πόρων που θα χορηγηθούν εκτός από το έμπολα Υπάρχουν και, και τρεις άλλες του επίπεδου κρίσης. Ιράκ, Συρία, Κέντρο Αφρική, Αφρικανική Δημοκρατία και Σουδάν, Νότιο Σουδάν. Όσοι είπατε ότι πρέπει να, να είμαστε περισσότερο ελαστικοί, να υπάρχει περισσότερη δημοσιονομική ευληγησία, γιατί μόνον η γρήγορη αντίδραση μπορεί να σώσει ζωές, Έχετε δίκιο, αλλά ελπίζω ότι η ελαστικότητα αυτή στην ανταπόκριση θα υπάρξει σύντομα σε έναν τέτοιο κόσμο με τέτοια με τόσο μεγάλα προβλήματα. Τώρα, πώς εξαπλώνεται ο ιός μέσω γοριλών, χιμπατζίδων, σκαντζοχύρων αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τον υπόλοιπο κόσμο διότι δεν βλέπουμε τέτοιου είδους κίνηση. Επομένως δεν υπάρχει παγκόσμιος κίνδυνος, έτσι μας λένε οι γιατροί. Η ελεύθερη διακίνηση, τα ταξίδια και ο τουρισμός είναι κίνδυνος ή όχι. Ίσως να μην γνωρίζετε κάτι. Οι γιατροί χωρίς σύνορα δεν συνάντησαν ούτε ένα κρούσμα στο προσωπικό τους και όμως ταξιδεύουν και είναι επιτόπου δηλαδή ο έμπολα είναι ελέγξιμος αν πλύνει κανείς τα χέρια του πριν να μπει σε αεροπλάνο ας πούμε και το φροντίζουν αυτό οι αεροπορικές εταιρείες. Υπάρχουν προληπτικά μέτρα λοιπόν και δεν πρέπει να ανησυχούμε ότι είναι επικίνδυνα τα ταξίδια και οι μετακινήσεις. Αντίθετα, αν δεν μπορούμε πια να στείλουμε και άλλους γιατρούς και να βγάλουμε από τις μολυσμένες περιοχές τον πληθυσμό, καθώς και νοσοκόμες και γιατρούς, τότε ακριβώς θα εξαπλωθεί περαιτέρω η μόλυνση. Όσο δεν την καταπολεμούμε τόσο ψηλότερος ο κίνδυνος να αλλάξει ο ιός και να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνος ε, προς στιγμήν υπάρχει ε, εφαρμόζουμε ό,τι υπάρχει από εμβόλια και άλλου είδους θεραπείες αλλά να είμαστε σωστοί έχουμε περιορισμένες ποσότητες από όλα αυτά θέλουμε να βοηθήσουμε τους πάντες αλλά δεν μπορούμε τουλάχιστον ακόμα και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταπολεμήσουμε τον έμπολα από την αρχή Τώρα το κάνουμε με όσο το δυνατόν επιθετικότερο τρόπο, στεναρότερο τρόπο. Τέλος για το συντονισμό. Συμφωνώ πολύ ότι ο συντονισμός σώζει ζωές. Έχουμε πολύ ισχυρό μηχανισμό συντονισμού από τον ΟΗΕ με τον Δόκτωρο Ναμπάρο και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αλλά επίσης πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς γιατί 28 χώρες μέλη συν την αν όλοι προσπαθούσαν μεμονωμένα να βοηθήσουν θα πίεζαν ε, χωρίς λόγο εκείνους που δρούν επιτόπου. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι σε θέση να σας πω, αν και ξέρω ότι πρέπει να τελειώνω, ότι πέρυσι με τη βοήθειά σας, με την υποστήριξή σας, οργανώσαμε το κέντρο συντονισμού που δίνει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να δράσει με μια ενιαία στάση όταν χρειάζεται. Το Συμβούλιο τώρα, ο κύριος Δελαβέντοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τον ιό αυτό σαν μια βασική προτεραιότητα. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επίτροπο Αγγιόγκεβα για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα και για τον ξεκάθαρο τρόπο με τον οποίο στις απαντήσεις της ξεκαθάρισε τις δράσεις που έχει αναλάβει. Σε λειτουργικό επίπεδο οι ανάγκες ε, επιτόπου είναι μεγάλες. Προσωπικό, ε, ιατρικό, εργαστηριακό, ανθρωπιστικό. Υπάρχουν και άλλες ανάγκες στον τομέα της υγιεινής, όχι της υγείας, λόγω ακριβώς της ε, διάλυσης ουσιαστικά των υπηρεσιών υγείας στη Λιβερία και στη Σιεραλεόν ελλείψεις σε φάρμακα, ελλείψεις σε τρόφιμα, ελλείψεις στη διοίκηση, ελλείψεις στην ασφάλεια. Όλα αυτά κινδυνεύουν στο να τονίσουν την ε, εξάπλωση του ιού αυτού θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των αφρικανικών χωρών, ιδιαίτερα αυτών που είναι ιδιαίτερως εκτεθειμένες. Την προηγούμενη εβδομάδα, στα πλαίσια της συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, μάλλον την επόμενη εβδομάδα, θα συζητήσουν και θα συντονίσουν τις περαιτέρω απαντήσεις στην κρίση. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πλαίσιο λειτουργικό απάντησης που καλύπτει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απειλές διασυνοριακού τύπου. Οι υπηρεσίες υγείας και υγιεινής των κρατών μελών είναι σε θέση ε, να κρίνουν την πιθανότητα άφηξης ασθενούντος από τον ιό στην Ευρώπη. Κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε να προετοιμαστούν σωστά για μια τέτοια έλευση αν και ο κίνδυνος για να κολλήσουν την ασθένεια ε, αυτοί που συνταξιδεύουν θεωρείται ε, πάρα πολύ χαμηλός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το Συμβούλιο λοιπόν. Έχει κλείσει η συζήτηση. Πριν περάσουμε στην επόμενη συνάντηση, θα ήθελα να κλείσουμε το θέμα των πρακτικών στα γαλλικά. Εγώ ζήτησα να ελέγξουν οι υπηρεσίες ε, του Κοινοβουλίου την εφαρμογή του κανονισμού σε σχέση με τις τροπολογίες. Το άρθρο 192 λέγει στο σημείο του 3 εφόσον τα πρακτικά αμφισβητηθούν